Okay. Good afternoon. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ συχνά, ξέρετε, μας λείπει χρόνος, γι' αυτό προτείνω να αρχίσουμε αμέσως. Δεδομένων και όλων των ε, θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια. Σήμερα το πρωί η μερίσια διάταξη της συνεδρίασής μας άλλαξε κάπως, γι' αυτό θα αρχίσουμε με το σημείο 14 την έκθεση για το διαδίκτυο και τις αγορές ναρκωτικών. Θα έχουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Κόστελ, διευθυντή του EMCDDA και από έναν πρόσωπο της Europol, το κύριο Βασιλάουσκας. Θα ήθελα επίσης και να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, κάνει μερικά πρόσθετα σχόλια. Ίσως θυμάστε ότι στις 5 Απριλίου και οι δύο οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συντάξουν την δεύτερη ετήσια έκθεση για τις ε, αγορές ναρκωτικών για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ε, διαδικτυακό εμπόριο ναρκωτικών, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τρίτες χώρες, για τους ερευνητές και για εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της βιομηχανίας και διάφορων εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει προς το παρόν και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόστελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σήμερα θα σας παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αγορά Ναρκωτικών. Δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη ε, με τον, ε, από τον Επίτροπο κ. Βραμόπουλο και τον ε, Διευθυντή της Ευρωπόλη, τον συνάδελφό μου. Η έκθεση αυτή είναι βασισμένη σε μια σύνθεση πληροφοριών και συνεισφορέ εμπειρογνωμόνων, στατιστικών στοιχείων και πληροφορίες που είναι διαθέσιμε από την παρακολούθηση της κατάστασης σχετικά με τις αγορές ναρκωτικών και σε συνεργασία με τις ε, εθνικές αρχές. Αυτό καθιστά και μοναδική την έκθεση, δηλαδή υπάρχει μια στρατηγική ανάλυση η οποία γίνεται δυνατή μόνο με τον συνδυασμό δεδομένων πληροφοριών που προέρχονται από δύο διαφορετικούς ε, κόσμους οι οποίοι συνήθως δεν συνεργάζονται. Από την ε, από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτηση και της μείωσης αυτής. Τι έχει αλλάξει από την πρώτη έκθεση πριν από τρία χρόνια και ποιες είναι οι καινούργιε γνώσεις που έχουμε μετά από τη συνεργασία με την Ευρωπόλη και τους υπόλοιπους εταίρους. Αυτό θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Καταρχάς, για πρώτη φορά έχουμε μια εκτίμηση του όγκου της ε, κίνησης του εμπορίου, και του εμπορίου ναρκωτικών. Περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, κοστίζει το εμπόριο ναρκωτικών. Υπάρχει μια εκτίμηση περίπου από 21 έως 31 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι η πρώτη φορά που η εκτίμηση αυτή έχει βασιστεί σε δεδομένα τα οποία έχουν, έχουμε συλλέξει από όλη την επικράτεια της Ένωσης. Ε, δεδομένα για παράδειγμα που συλλέγουμε από τους χρήστες που βρίσκονται σε προγράμματα αποτοξίνωσης και προσπαθούμε όσο περνά ο καιρός να βελτιώνουμε το σύστημα συλλογής δεδομένων έτσι ώστε η εκτίμηση να είναι πιο κοντά στα πραγματικά όσα Εκτιμούμε ότι ίσως ε, να είναι ακόμα περισσότερο, περισσότερα τα έσοδα, ακόμα υψηλότερο το ποσό από το, την αγορά ναρκωτικών. Το μερίδιο της αγοράς για κάθε μία από τις ναρκωτικές ουσίες έχει ως εξής 38% από την κάναβη, 28% ε, για ηρωίνη, 24% για κοκαίνη και μετά αλλάζουμε κατηγορία ναρκωτικών. Περνάμε στη, τα ναρκωτικά με το χαμηλότερο μερίδιο, 8% για διάφορες αμφεταμίνες και 3% για έκσταση MDMA. Τώρα θα με ρωτήσετε και τι γίνεται όμως με το NPS. Ο οργανισμός μας και η Ευρωπόλ έχουν ασχοληθεί με το θέμα των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, τα οποία πολλούνται νόμιμα ως ε, αντικατάσταση παράνομων ουσιών. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι ο αριθμός, η διαθεσιμότητα των ε, ουσιών αυτών ε, φαίνεται να μην μειώνεται. Πέρυσι, μαζί με την Ευρωπόλ, εντοπίσαμε 100 νέες ουσίες, οι οποίες ε, εμφανίζονταν πρώτη φορά. Επίσης, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο συντονίζουμε, αυτή τη στιγμή παρακολουθεί 560 τέτοιες ουσίες, 70% των οποίων έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση και να αναφερθώ στο τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο αντίκτυπος και πώς θα επηρεάσει το νόγκο εργασία στο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Το θέμα δεν είναι να εντοπίσουμε μόνο τις νέες ουσίες, αλλά να συνεχίσουμε τον έλεγχο για το αν θα εμφανιστούν ξανά και το τι γίνεται, πώς ε, κάνουν τον κύκλο τους αυτές οι ουσίες. Είναι λοιπόν μια μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, το οποίο βέβαια σημαίνει και αυξημένο διοικητικό φόρτο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για κάθε μία από τις ουσίες αυτές ή και τις ομάδες ουσιών αυτών, η έκθεση παρουσιάζει μία περιεκτική ανάλυση της κατάστασης και προτείνει διάφορους ε, τρόπους ε, δράσης σε συνεργασία πάντα με την Ευρωπόλ και βασιζόμαστε στην πρώτη έκθεση για τις ε, αγορές ναρκωτικών. Στην έκθεση αναφέρονται τέσσερις τρόποι με τους οποίους επηρεάζουν τα ναρκωτικά την κοινωνία. Ο πρώτος είναι ο σύνδεσμος με α... Ε, η σύνδεση μάλλον με άλλες μορφές εγκληματικότητας. Δεύτερον, ο αντίκτυπος ε, στην νόμιμη οικονομία, τρίτον η διαφθορά κυβερνητικών οργανισμών και τέταρτον το οποίο δεν είναι λιγότερο σημαντικό είναι οι αρνητικέ επιπτώσεις ε, που έχουν στην κοινωνία με ευρύτερη έννοια, δηλαδή ε, έγκλημα και βία που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, περιβαλλοντική καταστροφή, αντίκτυπο στην οικογένεια και στην ε, κοινωνία. Επίσης προσπαθούμε να αναλύσουμε τις εξελίξεις και το τι προκαλεί τις αυξήσεις στην αγορά των ναρκωτικών και ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις εκεί. Έπειτα, όπως παρουσίασε και ο Επίτροπος κ. Ευραμόπουλος, ε, ασχολούμαστε με το ρόλο που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην αγορά ναρκωτικών, παρέχοντας δηλαδή και ε, ευκαιρίες πώλησης, αλλά και ευκαιρίες μείωσης ε, της πώλησης. Αναφέρεται λοιπόν και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η αγορά των ναρκωτικών έχει κινητήριους μοχλούς το κέρδος και την εξουσία. Και ο αντίκτυπο που έχουν τα ναρκωτικά στην κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αν θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση τους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέες στρατηγικές έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ε, υγεία και η ευημερία των πολιτών μας. Τέλος, αναγνωρίζουμε ότι το όλο σκεπτικό πίσω από την αγορά ναρκωτικών είναι ότι η προσφορά έχει διαδραστικό ε, ρόλο με την ζήτηση. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν με επιτυχία τις αρνητικές συνέπειες ε, της χρήσης ναρκωτικών και για τους χρήστες αλλά και για την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία σε όλες τις επιτυχίες αντιμετώπισης, δηλαδή στην αποτοξίνωση, στην ψυχολογική υποστήριξη, στην καταπολέμηση, ε, στη σύλληψη των ε, δραστών κτλ. Τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση ε, στο ρυθμό αλλαγής της αγοράς. Έχουμε ολοένα και γρηγορότερα μεταβαλλόμενες τεχνικές αυξανόμενη πρόοδο στην τεχνολογία και αύξηση της εγκληματικότητας στην Ευρώπη. Έχουν διαπιστωθεί νέες επιθετικές στρατηγικές και χρήση του διαδικτύου για προώθηση των ναρκωτικών ουσιών και για τη δημιουργία νέων χρηστών τα τελευταία χρόνια. Σήμερα Έχουμε ε, διάφορες προτεραιότητες ε, στην Ευρώπη. Τρομοκρατία. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν μαζική μετανάστευση. Αυξανόμενη αστάθεια και εμπόλεμε ζώνες πολύ κοντά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε για παράδειγμα τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία, στην Συρία, στον Νότιο Κάφκασο, στην Υποσαχάρη Αφρική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν τις ε, ιδανικές συνθήκες που απειλούν την επιτυχία της ε, πολιτικής μας κατά των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση αυτή είναι μια τόσο ε, σημαντική και επίκαιρη έκθεση. Πρέπει να μην χάνουμε την προσοχή μας, να μην στρέφουμε την προσοχή μας αλλού, αλλά αντιθέτως να δώσουμε μεγάλη προσοχή και να μην ξεχνάμε το ρόλο των ε, εμπλεκόμενων φορέων. Μαζί με την Ευρωπόλ και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη θα καταφέρουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Σας ευχαριστούμε. Αναφέρετε όχι μόνο τον αντικτύπο της χρήσης ναρκωτικών ε, στην κοινωνία και στο άτομο, αλλά και τη διασύνδεση με τις άλλες μορφές εγκλήματος. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο παρά αυτά στον κύριο Βασιλάους από την Europol. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λαθρεμπόριο και η λαθρεία παραγωγή ναρκωτικών αποτελεί ε, μία από τις πιο καινοτομικές αγορές και τις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές στην Ευρώπη είναι πολύ περίπλοκη και έχει και διασυνδέσεις με άλλες μορφές εγκλήματος, μεταξύ άλλων και με την τρομοκρατία και αποτελεί βασική απειλή λοιπόν για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρθηκε από τον επικεφαλής, η εκτιμήσεις μας είναι 45 δισεκατομμύρια ανά έτος. Και αυτό μάλιστα έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις για το 2014. Έχουμε και επιπρόσθετες ε, ε, επιβαρύνσεις ε, και ενδεχομένως λοιπόν να είναι πολύ σε αυτό το ποσό, σε αυτό το αριθμητικό στοιχείο. Θα συνεχίσουμε όμως ε, να το αναλύουμε για τα επόμενα χρόνια. Η εκτίμηση της Europol είναι ότι έχουμε πάνω από 3.000 ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες δραστηριοποιούνται την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τρίτο ε, αυτών ε, με έναν ή μάλλον τρόπο ε, εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ένα τρίτο, δύο τρίτα εμπλέκονται στα πολυναρκωτικά. Δηλαδή με μια μεγάλη ποικιλία ναρκωτικών και λειτουργούν σε πολλαπλές χώρες και τομείς. Δεν τίθεται θέμα εθνικότητας ή εξειδίκευσης. Ε, μπορούν να δρουν ε, διασυνοριακά με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελεγχιστοποίηση του κινδύνου. Και οι οργανωμένες αυτές ομάδες ε, έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογή ό,τι φορά τις δραστηριότητε τους και τα μέλη τους. Έχουμε καλά, καλοργανωμένο δίκτυα, αλλά έχουμε και μικρά περιφερειακά δίκτυα που διανέμουν σε περιφερειακό επίπεδο τα ναρκωτικά. Χρησιμοποιούν επίσης ε, οδούς μεταφοράς και υποδομές, ε, ε, το Ροτοντάμ, το Αμβούργο, μεγάλους λιμένες, και καθημερινά καταφτάνουν τέτοιες ποσότητες ναρκωτικών σε μεγάλες αποστολές και επίσης και σε πακέτα. Είδαμε επίσης αύξηση στις θαλάσσιες μεταφορές με χαμηλότερο κόστος και επικοινωνιών και μεταφορών και αυτό ασφαλώς σημαίνει πιο αποτελεσματική έχει επιτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα και μεγαλύτερο κέρδος για αυτούς που εμπλέκονται. Εξακολουθούν να είναι μεγάλη ποικιλία στις ε, αγορές ναρκωτικών. Υπάρχουν κάποιες ε, σταθερές ε, δίωδοι για την διακίνηση που εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά υπάρχουν και καινούργιες τέτοιες οδοί. Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία, η από την Νοτιοαφρική προς την Ευρώπη, για παράδειγμα, η παραγωγή ναρκωτικών λαμβάνει η χώρα πιο κοντά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους καταναλωτές και αυτό ισχύει κυρίως για την Κάναδα και τα σχετικά ναρκωτικά. Και η παγκοσμιοποίηση διευκολύνει την ανταλλαγή και νόχαου και τεχνογνωσίας και γνώσης. Επίσης μπορεί κανείς ε, από το διαδίκτυο να δει πώς μπορεί να χτίσει μία επιχειρήση από το μηδέν. Επίσης ε, η... το εμπόριο ναρκωτικών στο διαδίκτυο αυξάνεται διαρκώς. Και παρά το γεγονός ότι το dark web, το σκοτεινό δίκτυο, καταπολεμείται από τις αρχές επιβολής του δικαίου, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οδός σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με την τρομοκρατία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν συστηματικοί σύνδεσμοι συνδέσεις μεταξύ τρομοκρατίας και ελαττρομπορίου ναρκωτικών, ωστόσο υπάρχουν τέτοιες συνδέσεις, αρκετά ευκαιριακές αν θέλετε. Στην Europol έχουμε διαπιστώσει υποθέσεις που συνδέονται κυρίως με τα ιστορικά στοιχεία για τους ε, αλλοδαπούς μάχητες. Λάβαμε σχετικά στοιχεία πριν από κάποιο καιρό, αλλά όπως σας είπα δεν είναι συστηματική αυτή η σχέση. Δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστον επί του παρόντος. Στην επόμενη διαφάνεια ε, βλέπετε την διακίνηση για την ε, Κάνοβη. Ολλανδικής και Βιετναμεζικής ε, παραγωγής κυρίως. Ε, δίδεται και χορηγείται τεχνογνωσία για να πώς να για παράδειγμα τα επίπεδα THC. Και η καλλιέργεια συνδέεται και με τη βία μεταξύ των σχετικών ομάδων. Συνδέεται και με εμπορία ανθρώπων και σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική καλλιέργεια της κάναβης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το cannabis ε, resin, το βλέπετε ποιες είναι οι, οι από κάναβη, βλέπετε ποιες είναι οι οδοί. βλέπετε πώς είναι η διακίνηση προς τις χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια πρόσφατη, Ενδεχομένω σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη ρητίνη από Κάναδη από το Μαρόκο είναι η χρήση πλοίων που μεταφέρουν την Κάναβη ανατολικά τη Μεσογείου προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής όπου φυσικά υπάρχουν και ασταθή περιβάλλοντα τα οποία ε, υπόκειται εκμετάλλευση. Το Δεκέμβριο του προσμένου έτου του 2015 η Europol υποστήριξε τις Ιταλικές Αρχές σε μια επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση πάνω από 14, από 14, σε 14 τόνους ε, κάναβης με, σε ένα πλοίο ε, με σήμερα του Παναμά και υποστηρίχθηκε από τις Ισπανικές και τις Ελληνικές Αρχές η επιχείρηση αυτή αυτό αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα τέτοιων συλλήψεων και κατασχέσεων σημαντικού όγκου κάναβης στη Μεσόγειο. Από πέρσι τον Ιούνιο έχουμε κατασχέσει πάνω από 60 τόνους κάναβης. Και 100 κιλά και περισσότερο κοκαίνης. Πρόσκειται λοιπόν για δίκτυα τα οποία λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Άρα όλες αυτές οι ενέργειες έλαβαν χώρα υπό ε, συντονισμό διεθνή και η όλα συνέδραμε. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τη ηρωίνης. Η διαφορά είναι ότι οι μεγάλες αποστολές φτάνουν στην Ευρώπη και ε, έχουμε όλο και πιο πολλές κατασχέσεις. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι βλέπουμε όλο και πιο μεγάλες αποστολές, μεγάλου όγκου, 100 κιλά ηρωίνης και πάνω. Και ακόμα και τόνους, δύο τόνους την προηγούμενη εβδομάδα, στην, ε, την μήνα στην Ελλάδα, ένα τόνο στην Ολλανδία. Οι μεγάλες, μιλάμε λοιπόν για μεγάλους, ε, μεγάλες ποσότητες οι οποίες εντοπίζονται. Και βλέπετε πέρα από την παραδοσιακή οδό των Βαλκανίων έχουμε τον Νότιο Κάφκασο, τη Συρία, το Ιράκ ω άλλη εδώ Και επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία παραμένει η βασική πύλη για την ηρωίνη, την εισαγωγή ηρωίνης ε, στην Ευρώπη. για την παραγωγή τώρα στην, στη στην Ευρώπη. Έχουμε συνδράμει στα μελη για την εντοπισμό εργαστηρίων που μετατρέπαν την, ε, ε, τη μορφή σε ηρωίνη, στην Ισπανία για παράδειγμα. Οι τουρκικές ε, και πακιστανικές ε, και αλβανικές επίσης ομάδες είναι ευθύνονται για μεγάλο τμήμα των ε, εισαγωγών. Για την κοκαίνη δεν θα σας περιγράψω ε, το διάγραμμα, το βλέπετε άλλωστε στη διαφάνεια με χρωματική επισήμανση και βλέπετε λοιπόν πως από πού προέρχονται από την Κολομπία, τη Βραζιλία, και την Βενεζουέλα. Στην Κεντρική Αμερική ε, είναι βασική περιοχή διέλευσης των ε, αποστολών αυτών προς την ε, Ευρώπη. Κάτι άλλο καινούριο. Πέρα, α, μάλλον ότι πλέον χρησιμοποιούνται και οι οδοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως τώρα για άλλα ναρκωτικά πλέον και για κοκαίνη. Από Μαρόκο, για παράδειγμα, προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτά τα δίκτυα, λοιπόν, παρέχουν πλέον υπηρεσίες και υποστηρίζουν ε, το λατρεμπόριο κοκαίνης. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την εισαγωγή όγια στην Ευρώπη είναι σαφής νομίζω η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα σημεία εισόδου. Χρησιμοποιούνται διάφορες ε, μέθοδοι ε, αεροπορικά, μέσω τυχεδρομείων, ε, μέσω ιδιωτικών αεροπλάνων και μέσω κοντέινερ εμποροκυμάτων και βοτήγων μέσω θαλάσσης. Άμστερνταμ και Αμβέρσα είναι τα βασικά λιμάνια όπου καταφτάνουν οι αποστολές κοκαίνης, καθώς και τα μεγάλα λιμάνια όλης της Δυτικής Ευρώπης που αποτελούν στόχο για το οργανωμένο έγκλημα, όπου χρειάζεται χημική εξαγωγή χημική επεξεργασία έχουμε επίσης ε, σημειώσει κάποια ζητήματα και βλέπετε ποιες είναι επίσης οι τάσεις και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και φυσικά τίθεται θέμα ε, σε, μεγάλες, σε πολλές περιπτώσεις διεφθαρμένων λιμενικών. Είναι μεγαλύτερο το πεδίο λειτουργίας των ε, λαθρεμπόρων κοκαίνης, αλλά εξακολουθούν να υπηρεσχύουν οι Κολομβιανοί και οι Ιταλοί έχουμε και ομάδες από την Ολλανδία ε, και την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πιο σημαντική εξακολουθεί να είναι από, το, από, το, από την Ισπανία και την Ολλανδία. Οι οργανωμένες ε, ομάδες ε, οργανωμένου κλίματος από τα Βαλκάνια αποτελούν επίσης μεγάλη απειλή σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο κοκαίνης εγκαθίστανται και σε διάφορες ε, και σε άλλες χώρες, σε χώρες ε, ε, παραγωγής στην Νότια Αμερική ή σε χώρες διαμετακόμισης, στην Νότια Αφρική για παράδειγμα και έτσι μπορούν να διευκολύνουν και να συντονίζουν τις επιχειρήσεις. Βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια τα διάφορους, διάφορους τρόπους λατρεμπορίου κοκαίνης. Βλέπετε εδώ πέρα για ένα το ξύλο και, ότι, και τις, τα κενά που υπάρχουν εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του εμπορευματικού εμπορευματοκιβετίου και κατασχέθησαν πάνω από 100 κιλά κοκαίνης. Χρησιμοποιήθηκε διπλό μόντους operandi ίσως να χρησιμοποιηθεί και το ίδιο κοντέινερ από δύο διαφορετικά δίκτυα κυκλώματα. Ίσως και από ένα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για σύμπτωση ή για κάτι καινούριο, ένα νέο τρόπο λειτουργία. Πάντω σε κάθε περίπτωση θα το παρακολουθήσουμε. Συμφωτικά, ναρκωτικά. Παράγονται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζεται αυτό. Τα πιο πολλά καταναλώνονται άλλωστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον τα πιο πολλά ευρωπαϊκής παραγωγής καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό οδηγεί σε, σε σημαντικό εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε στο χάρτη στα αριστερά την ε, ανακάλυψη παράνομων εργαστηρίων τέτοιων ναρκωτικών βάσει το, της συλλογής δεδομένων που συλλέξαμε και βάσει των δεδομένων που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη. Βλέπετε όμως ε, τη συγκέντρωση τέτοιων εργαστηρίων για την παραγωγή συμβατικών ναρκωτικών. Δεν θα σας ε, αναλύσω τη διαφάνεια αυτή και πάμε κατευθείαν στην επόμενη. Σε ό,τι αφορά τα συμφετικά ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε Ολλανδικέ, Γερμανικέ, Βρετανικέ και Βέλγικε ομάδε οι οποίε δρούν στον τομέα αυτό. Και σε ό,τι αφορά το MDMA και την σαφαταμίνη, όλο ιδιαίτερω. Και επίση βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες είναι υπεύθυνε και για τη διανομή και βλέπουμε ότι υπάρχει διασύνδεση με την καναβή και την κοκαίνη. Ενώ οι βιετναμέζικες ομάδες που διαδραστηριοποιούνται για παράδειγμα στην ε, στις αμφεταμίνες ε, δραστηριοποιούνται και στις, ε, στο εμπόριο κάναβης. Αυτά τόνου BMK κατασχέθησαν στην Πολωνία πέρσι. Συλλάβαμε έναν Πολωνό υπήκονο, υπήκο, και δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά οι 7 τόνοι σε BMK αποτελούν σημαντικό ποσό, σημαντικό όγκο. Οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες τώρα αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην στη διαβάσω το κείμενο, να σας πω δύο-τρία πράγματα επιγραμματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω για το ποιο είναι το όφελο των ψυχοτρόπων αυτών ουσιών για τα κυκλώματα. Και αυτό βασίστηκε σε μια υπόθεση στο Βέλγιο πριν από τρία χρόνια. Ανακαλύφθηκε λοιπόν ένα εργαστήριο παραγωγής ψυχοτρόπων ουσιών και η αστυνομία κατάσχεσε 285.000 πακέτα τέτοιων νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Ένα πακέτο κάνει περίπου 25 ευρώ και αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να βγάλετε αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαζόταν περίπου 350.000 επενδύσεις κάποιες δηλαδή επενδύσεις σε εξοπλισμό με 350.000 δηλαδή ευρώ μπορεί κανείς να βγάλει 7 εκατομμύρια Εδώ λοιπόν βλέπουμε τεράστιες ε, διαφορές και μεγάλο όφελος προφανώς για τους εγκληματίες. Στην επόμενη διαφάνεια θα βρείτε το τελευταίο παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, το εμπόριο στο διαδίκτυο. Μια επιχείρηση η οποία διεξήχθη στην Ουγγαρία πριν από τέσσερα χρόνια. συνελήφθη σε ένα άτομο πριν από τέσσερα χρόνια γιατί πολλούς MPS ε, στο τη διακριτική σελίδα. Πουλούσε περίπου 100 μονάδες ανά εβδομάδα. Αλλά συνελήφθησε, έκλεισε το κατάστημα και δύο χρόνια αργότερα πάλι λειτουργούσε η ιστοσελίδα, ε, ενώ κρατούταν ακόμα ο υπεύθυνο και προέκυψε ότι οι νέοι πάροχοι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον προηγούμενο, αλλά χρησιμοποιούσαν το όνομα το οποίο ήταν ήδη γνωστό στους πελάτες τους. Οι Ουγγρικές Αρχές λοιπόν, με την υποστήριξη και κάποιων άλλων κρατών μελών και της Europol, ε, ανακάλυψαν και εξάρτησαν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονταν πίσω από την ιστοσελίδα αυτή, αλλά και από άλλες πολλές ιστοσελίδες με παρόμοιο τρόπο λειτουργίες, πολλούς φανουσίες από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια νέα επιχείρηση πρώην ανέργων ατόμων με με εκείνη ιστορία και με δομές τέτοιες. Προσπαθούμε λοιπόν να αποφεύγουμε τέτοιες ε, Προσπαθούσαν να αποφύγουν λοιπόν τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες που συμπεριλαμβανόντουσαν στις σχετικές λίστες. Εδώ βλέπετε και κάποιες εικόνες από άλλες τις ιστοσελίδες που λειτουργούσαν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τον Ιούνιο του 2015 ωστόσο πώλησαν Facebook tablets, νέα ψυχοτρόπους ουσία, και αυτό κατέληξε και οδήγησε 15 νέους στο νοσοκομείο σε μία νύχτα. Η ουσία αυτή, το Facebook Tablet, δεν ε, απαγορευόταν τότε. Έκαναν λοιπόν έρευνες οι αρχές για τους πελάτες, στους πελάτες ε, που είχαν χρησιμοποιήσει τέτοια προϊόντα και τελικά κατέληξα στη σύλληψη 6 ατόμων. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα συντομία της συγκεκριμένης επιχείρησης της οποίας ηγήθηκε η Ουγγαρία και υποστηριχθήκε από την Europol και από άλλες χώρες. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε αυτές τις εκθέσεις και κυρίως τον αριθμό 560 ουσίες είναι στην αγορά. Και σκέφτομαι τι ωραία που ήταν όταν μιλούσαμε μόνο για τσιγάρα και αϊνόπνευμα. Δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς όλες αυτές τις νέες ουσίες. Ε, δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει κάτι να προσθέσει για αυτό το θέμα. Όχι απαραίτητα. Οπότε θα ρωτήσω αν ο κύριος Μπόνι θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτής της ε, περιστατωμένης έρευνας. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλό παράδειγμα καρποφόρα συνεργασίας ανάμεσα ε, ευρωπαϊκά, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς. Είναι καλή έκθεση αυτή ο σημείο αναφοράς ε, για την Europol, την Κομισιόν και όλους μας. αλλά και για την ε, MCDDA ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, αλλά και όσον αφορά πολιτικές που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ποιες είναι οι προκλήσεις όπως εσείς μας αναφέρατε. Πρώτον, η αύξηση ε, του οικοσυστήματος, δηλαδή παραγωγή, διακίνηση, πώληση. Για ότι βλέπουμε ότι ορισμένε ομάδε οργανωμένου εγκλήματο ε, φτιάχνουν νέε μορφέ συμμαχιών ανάμεσα σε, που, που ξεπερνούν τα εθνικά και γεωγραφικά σύνορα. Ο οικονομικός αντίκτυπο, όπω υπόθηκε, αυξάνεται με, τον αρνητικό, με αρνητικό τρόπο καθώς η αξία της αγοράς ναρκωτικών εκτιμάται στο επίπεδο των 21 με 31 δι ευρώ ετησίως. Δεύτερο σημείο είναι η συγκέντρωση σε έναν ε, συγκεκριμένο αριθμό θεσπισμένων αλλά και αναδυόμενων ε, περιοχών ε, στην Ευρώπη με ειδικευμένες διόδους για την διακίνηση των ναρκωτικών νέες και αναδυόμενες ζώνες παραγωγής σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ε, το παράδειγμα της παγκοσμιοποίησης δηλαδή της ε, αλυσίδας, της εγκληματικής αλυσίδας των ναρκωτικών. Είναι σαφές πως και το ίντερνετ δημιουργεί νέες δυνατότητες προώθησης ε, των ναρκωτικών αλλά και Διάδοση των γνώσεων για το πώς να τα χρησιμοποιήσει κανείς και πώς να τα αποκτήσει. Ο ρόλος δε του Darknet αυξάνεται επίσης. Τρίτο σημείο είναι η πολυδιάστατη, ο πολυδιάστατος αντίκτυπος των μεγεθυνόμενων αγορών ναρκωτικών και ευκολότερη πρόσβαση στα ναρκωτικά, ιδιαίτερα στα νέα ναρκωτικά, όπως οι νέες ψυχο ε, ε, τρόπες ουσίες. Ο αντίκτυπος αυτός είναι πολύ επιζήμιος για την οικονομία, για την υγεία των ανθρώπων, για το 1% των Ευρωπαίων ε, ενηλίκων χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά σε καθημερινή βάση. Σημαίνει αυτό 6 εκατομμύρια κόσμος. Και επίσης αυτό προσθέτει στην ε, ριζοσπαστικοποίηση κοινωνικών ε, συμπεριφορών σε ορισμένες χώρες. Τίθενται επίσης ε, ερωτήματα όσον αφορά την προφανή σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη της αγοράς των ναρκωτικών και των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, γιατί σαφώς υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη διακίνηση ναρκωτικών και τις, τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Περιγραφή της αγοράς και χωρίς της αγοράς πρέπει να εστιάσουμε στην συστηματική ανάλυση και την πρόγνωση, πρόβλεψη ε, της επιχειρηματικότητας, τα νέα, τους νέους τρόπους χρήσης των ναρκωτικών, επίσης τους νέους κινδύνους για τους ανθρώπους λόγω της νέας σύστασης των ε, ναρκωτικών, πράγμα που είναι κλειδί για επιχειρησιακού ε, λόγους. Επίσης, είναι δραστήρια συμμετοχή όλων των θεσμών που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, το ρόλο δηλαδή των σημείων εστίας αλλά και ε, των κόμβων αλλά και της MCDDA. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ευρωπαϊκή συνεργασία για να αναπτυχθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και στεναρές και γρήγορες παρεμβάσεις ώστε να μπλοκάρετε η πρόσβαση στα ναρκωτικά και στα ψυχοτρόπες ουσίες. Ξέρουμε πως δεν είναι εύκολο, ότι υπάρχουν πολλά κρίσιμα σημεία, υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά και συνεργασία που γίνεται ανάμεσα στα κρατημέλη για τις νέες λύσεις σε σχέση με τις ψυχοτρόπες ουσίες και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια η έλλειψη συντονισμού μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους κάθε είδους. Χρειάζονται ισορροπημένες πολιτικές ώστε να μειωθεί η παροχή, η προμήθεια σε ναρκωτικά και βοήθεια βέβαια προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ναρκωτικά. Εκεί είναι ο τομέας των πολιτικών δημόσιας υγείας. Θα ήταν καλό από καινούργου καιρό να οργανώνεται κοινή συνεδρίαση ανάμεσα στην Επιτροπή μας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος που εντός των αρμοδιοτήτων της είναι και η υγεία και η δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να, ζητήσω, να ρωτήσω τον κύριο Κούσδηλ τι είδου δυνατότητε, έχει ή χρειάζεται το κέντρο ε, MCDDA για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην, ε, στο ρόλο σχηματισμού πολιτικών. Ε, το νέο πλαίσιο για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό απαραίτητο και πώς μπορούμε καλύτερα να χειριστούμε το αυξανόμενο πρόβλημα των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί περιέχουν γιατί είναι ακόμα άγνωστες οι επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ουσιών. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν μόνο δήλωση αυτή που κάνατε, αλλά και ε, θίξατε πολλά ερωτήματα και σκέφτομαι τα νούμερα που ακούσαμε, ότι μπορεί κανείς δηλαδή να κερδίσει 24 δις ευρώ. Θυμάμαι ότι είχαμε προβλήματα να βρούμε 6 δις ευρώ για τη συμφωνία με την Τουρκία. Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς. Πάντως νομίζω ο συνάδελφος ε, θα μπορούσε να απαντήσει από την Europol. Όταν δούμε αυτές τις διαφανείς βλέπουμε διαφόρων ειδών ναρκωτικά αλλά και διαφορετικούς τρόπους ε, διακίνησής τους τόσο για να φτάσουν αυτά στην Ένωση όσο και για να διανεμηθούν εδώ. Οι δρόμοι που ακολουθούνται αλλάζουν συχνά, πράγμα το οποίο θα, βέβαια θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ίσως θα μπορούσατε κάτι να προσθέσετε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μπόνι για τα θετικά του σχόλια. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και γενικότερα αυτήν την Επιτροπή για την συνεχιζόμενη στήριξη που δείχνει στο έργο μας. Τώρα, συγκεκριμένα για την ερώτησή σας για τα μέσα και για τους πόρους που ε, είναι διαθέσιμοι. Υπάρχει μια νέα νομοθεσία που προετοιμάζουμε σχετικά με την προσέγγιση που θα εθετήσουμε για τις νέες ε, ψυχοτραστικές ουσίες. Αυτή τη στιγμή προβλέπονται τρία στάδια. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μετά εκτίμηση κινδύνου και μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο των ουσιών αυτών. Αν δεν κάνω λάθος, χθες η Κορεπέρα έλαβε μία απόφαση για μία αναθεώρηση, περιορισμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας. Αλλά πιστεύω πως το κεντρικό, ε, πιο σημαντικό σημείο είναι τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η τροποποιημένη πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού δεν θα είναι αρκετή, πιστεύω, οποιαδήποτε τροποποίηση για να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις που έχουν προκύψει και πιστεύω ότι δεδομένου τούτου έχουμε την ίδια άποψη με την Επιτροπή σας. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε και όλα στο στάδιο των προτάσεων, θα ήθελα να έχω και τη δική σας συνεισφορά για το τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τους πόρους χρειάζονται σίγουρα πρόσθετη πόρη έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον αντίκτυπο αυτής της αυξανόμενης χρήσης ε, ναρκωτικών ουσιών. Και είμαι πεπισμένο ότι θα βρούμε στο τέλος κάποια λύση, διότι ξέρω ότι η Κομισιόν έχει δείξει ισχυρή δέσμευση, αλλά και ε, το Συμβούλιο έχει κάνει υποσχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως εφόσον υπάρχει η βούληση θα ε, έχουμε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αυξήσουμε τους πόρους που χρειάζονται για την καταπολέμηση των, ε, της αύξησης των ε, χρήστες συναρκωτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα πάρα πολλές υπηρεσίες ζητούν αύξηση των κονδυλίων και όχι μόνο εσείς, αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση όντως. Κύριε Βασιλέως Κασά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σε σχέση με την αλλαγή των δρομών ε, που χρησιμοποιούνται, με την διαφοροποίηση, όπως είδατε και από τα βέλη στις διαφάνειες, ε, υπάρχουν διάφορες τάσεις, διάφορες ενδείξεις που ε, έχουμε συλλέξει από συγκεκριμένες περιπτώσεις, από έρευνες. Έχουμε δει λοιπόν ότι έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, έχουν αλλάξει οι οδοί που χρησιμοποιούνται όμως οι ροές παραμένουν σταθερές, δηλαδή ε, εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου, υπάρχουν όμως διάφορες δυνατότητες αντιμετώπισης. Πράγματι υπάρχει διαφοροποίηση μεθόδων, διαφοροποίηση των ε, οδών που χρησιμοποιούνται, όμως αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ανέκαθεν άλλαζαν. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, αξιότιμους προσκεκλημένους, γιατί πιστεύω ότι κάναμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε και ενημερωθήκαμε για την κατάσταση. Σίγουρα η μάχη ε, δεν είναι εύκολη, όμως υπάρχει, υπάρχει ενημέρωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μια παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας και των ερευνητικών εργασιών. Θα ακολουθήσουν τρεις παρουσιάσεις που είναι όλες εξίσου χρήσιμες για την συζήτηση. Καταρχάς, μια παρουσίαση για την εξελόγηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που διεξήχθη από τη δική μας ε, ομάδα μελετών του Κοινοβουλίου και δύο μελέτες εμπειρογνωμόνων που αναθέσαμε για το θέμα αυτό. Αυτές οι μελέτες διεξήχθησαν για να στηρίξουν την έκθεση της Επιτροπής μας σχετικά με την ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία, κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης μάλλον έχει εισηγήτρια την κυρία Ιντφελ και βρίσκεται στη διάθεσή σας από χθες. Θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην ε, εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσει την ενδιάμεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω να σας παρουσιάσω την έκθεση. Όπως ε, είπατε και εσείς θα αρχίσω με τα θεμέλια πίσω, με το σκελετό αυτής της έκθεσης. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με το άρθρο 125 της συνθήκης, μας ζητήθηκε αυτή η έκθεση. Αυτή η έκθεση συνοδεύεται πάντα από την αξιολόγηση για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Προσπαθούμε δηλαδή να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα των προτάσεων που θα υποβάλει το Κοινοβούλιο στην έκθεση Ιδίας Πρωτοβουλίας. Αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, όπως ξέρετε, συνοδεύει την έκθεση της κυρίας Σίντφελτ και στόχο έχει να παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πλεονεκτήματα του ε, μηχανισμού ε, Δημοκρατίας Κρατούς και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όπως είπατε, είναι μια ενδιάμεση αξιολόγηση η οποία θα ολοκληρωθεί πριν την ε, δημοσίευση του σχεδίου έκθεση τη κυρία Σίνφελτ. Έχει λάβει υπόψη τα διάφορα γκρέφα εργασία τα οποία μα παρουσίασε η συγγήτρια και οι σκιώδεις και θα επικαιροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι μελέτε θα παρουσιαστούν από τον κύριο Μπάρντ, εξ μέρου τη ε, ΣΕΚ και τον κύριο ε, ΣΕΚ από την Μιλιά. η κυριότερη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στο σύστημα. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό ανάμεσα στην ε, δήλωση των αξιών που αναφέρονται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμόρφωση με αυτές στην πράξη από τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Τότε το κενό λοιπόν έχει κόστος οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Και οι αδυναμίες που έχουμε παρατηρήσει σχετίζονται καταρχάς με το πεδίο εφαρμογή της αρμοδιότητας, με την επιβολή των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ασάφεια σχετικά με τους ορισμούς. Συνεπώς υπάρχει μία ασάφεια στην διάκριση, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Υπάρχει δηλαδή ασάφεια στο ποιος κάνει τι στο θέμα επιβολής ε, του νόμου. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις στον συντονισμό των δράσεων. Τρίτον, οι φυστάμενοι μηχανισμοί έχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν αποτελεσματικότητας διότι δεν αντιμετωπίζουν απαρκώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου στην Ένωση. Τώρα, ποιες ε, είναι οι επιλογές που έχουμε νομοθετικές και μη έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος στο έγγραφο εργασίας, αλλά και εμπειρογνώμονες έχουν προτείνει να υπάρχει ένα διοργανικό σύμφωνο, το οποίο θα διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής, αλλά και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα ε, κράτη-μέλη της Ένωσης. Θα υπάρχουν δύο στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν αυτό το σύμφωνο. Καταρχά ετήσια επισκόπηση και παρακολούθηση του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ένα νέο δείκτη επιδόσεων. Από την άλλη, θα συμπεριλαμβάνει και ένα νέο κύκλο πολιτική, δηλαδή κάτι σαν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε σχέση τώρα με την ετήσια παρακολούθηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες πρωτού μπορεί αυτό να τεθεί σε ισχύ, κυρίως στο ε, πεδίο δράσης. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντολή να παρεμβαίνει έτσι ώστε να μπορεί να προστατεύσει τον συνταγματικό πυρήνα, δηλαδή τις αξίες που ε, διέπουν όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο είναι η νομική βάση μια τέτοια αιτήσια παρακολούθηση θα μπορούσε να βασίζεται στο άρθρο 352. Είναι η νομική βάση για τη δημιουργία της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το έργο της. Επίσης, το άρθρο 70. Άρθρο 70 αναφέρεται στα εσωτερικά και... εσωτερικές υποθέσεις και δικαστική συνεργασία. Ή το άρθρο 5, το οποίο αποτελεί τη νομική βάση για τις διοργανικές συμφωνίες. Θα μπορούσε επίσης να είναι και ένα συνδυασμός όλων των παραπάνω. Επίσης, υπάρχουν κάποιες ε, ερωτήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία, των ε, δίκτυ επιδόσεων, την κατανομή αρμοδιοτήτων στα θεσμικά όργανα και επίσης διάφορα προβλήματα σχετικά με την ε, δημοκρατία και τη λογοδοσία. Έπειτα ως προς το δεύτερο στοιχείο. Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, εδώ θα συμπεριλαμβάνεται και ετήσια ανταλλαγή απόψεων στα Εθνικά Κοινοβούλια, διακοινοβουλευτική συνεδρίαση, Βελτιώσει στο πλαίσιο για το κράτος δικαίου και μια δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ε, κινεί διαδικασίες επί παραβάση. Επίσης θα χρειαστεί και βελτίωση του ε, διαλόγου για το κράτος δικαίου μέσα στο Συμβούλιο. Χρειάζεται λοιπόν η εντολή για να γίνουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα προτείναμε ο κύκλος πολιτικής να συμπεριλαμβάνει και ένα σύστημα πρόβλεψης και αξιολόγησης της ευρωπαϊκής ανομοθεσίας στους τομείς αυτούς. Ταυτόχρονα, η διαδικασία προσχώρησης τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σύμφωνο των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, συνεχιστεί και να επισπευστεί. Έπειτα, κόστος, ε, σχέση όφελου των επιλογών πολιτική, Από ό,τι έχουμε δει στην επιστημονική βιβλιογραφία, ο ανεπαρκή έλεγχος της διαφθοράς, η έλλειψη θεσμικών ελέγχων, όλα αυτά έχουν αρνητικέ επιπτώσει σε πολλά επίπεδα ιδιαίτερα στις οικονομικές επιδόσεις. Σε μια πρόσφατη έκθεση σχετικά με το έγκλημα και τη διαφθορά φαίνεται ότι το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία ανέρχεται ε, από τα 218 στα 282 δισεκατομμύρια ετησίων. Επίσης, ε, χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και ας μην ξεχνάμε ότι κάθε πολίτης μπορεί να παίξει ρόλο. Εάν δεν υπάρχουν συνέπειες ε, στην παραβίαση νόμων, τότε θα μεταδοθεί στην κοινωνία η παραβατικότητα. Επίσης, ένα Τέτοιο σύστημα ελέγχου θα κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύκλος πολιτικής 7 εκατομμύρια. Και εφόσον βρεθούν οι κατάλληλοι και χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες συνέργειες θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισκόπηση αυτή και τι πληροφορίε αυτέ. Και τώρα θα δώσουμε παρά αυτό το λόγο στην κυρία συντόκτωρα Πέτρα Μπάρτ από το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης για να μας παρουσιάσει την ερευνητική εργασία του CEPS με τίτλο «Αξιολόγηση της ανάγκη των αναγκών και των δυνατοτήτων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σκόρμπορ για τη Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων». Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την ερευνητική εργασία και θα ήθελα να περάσουμε στη μεθεπόμενη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή και την ίδρυσή της είχε τις βασικές ε, αξίες της ε, γύρω από τις οποίες ε, θεμελιώθηκε και εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι βασικές και θεμελιώδεις αξίες. Έχουμε τρεις βάσεις οι οποίες και κατοχυρώνονται και στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κριτήρια της Κοπεχάγης δε εξασφαλίζουν ότι τα μελλοντικα κρατημέλη θα πληρούν τους όρους αυτούς προτού ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει όμως ε, ουσιαστικά κάποια μέθοδος παρακολούθησης της εφαρμογής των κριτηρίων αυτών μετά την προσχώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς έχει μηχανισμούς παρακολούθησης, οι οποίοι όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τότε που έχουν κατοχυρωθεί στις συνθήκες και όχι επειδή δεν υπήρχαν ε, Τέτοιε καταστάσεις όπου θα επιβαλόταν η χρήση της, του μηχανισμού αυτού, αλλά επειδή δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Και έτσι λοιπόν ε, η ακαδημαϊκοί κύκλοι ζήτησαν να υπάρξει μεταρρύθμιση σχετική. Μεταρρύθμιση από το Συμβούλιο, την ε, Επιτροπή, το Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν ε, βρίσκεται σε φάση δοκιμασίας μια σχετική διαδικασία. Φυσικά και υπάρχει κριτική. Γιατί το άρθρο 7.1 της συνθήκης θεωρείται ότι αποδυναμώνεται περαιτέρω. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίσουμε το ωφέλη της επισύνμασης του προβλήματος του κράτους δικαίου. Και έτσι περνάμε από την επικέντρωση στο άρθρο 7 σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στο ψήφισμα της 10ης Ιουνίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήλησε να υπάρξει ετήσια παρακολούθηση του κατά πόσο πληρούνται οι όροι αυτοί και να αναπτυχθούν κοινοί δείκτε. και η ομάδα μα που περιλαμβάνει και του καθηγητέ που κάθονται δίπλα μου εξέτασαν το ζήτημα αυτό. Βασικό λοιπόν σημείο αφετηρίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να θέσει στο στόχο του τα θέματα αυτά γιατί είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και επηρεάζεται ο Ευρωπαίος πολίτης πέρα από τα όρια του εθνικού κράτους μέλους. Και επηρεάζονται και οι πολίτες από άλλα κράτη-μέλη. Και επίσης από αυτό κρίνεται και η νομιμότητα και η νομιμοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει μηδέα αναγνώριση ε, των, της νομοθεσίας εάν δεν υπάρχουν τα κοινά αυτά πρότυπα πέρα από το α, και οικονομικό κόστος, η επικουρικότητα. φυσικά εξακολουθεί να ισχύει, δεν υπονομεύεται η συνταγματική αυτονομία των κρατών, αλλά δεν θα, ε, ο μηχανισμός αυτός δεν θα υπονόμευε την επικουρικότητα, ίσα ίσα θα την ενίσχυε. Άλλο σημείο αφετηρίας. Ε, το ε, Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μέσο, εξωτερικό μέσο, εξαγωγής της δημοκρατίας, όπου προστατεύεται ο πολίτης σε περίπτωση που υπάρχει θέμα αμφιβολίας. Αυτά τα κρατημέλη που βρίσκονται υποποίηση ασφαλώς θα α, επιτεθούν κατά της κριτικής. Θα κατηγορήσουν δηλαδή όσους ασκούν κριτική για προκαταλήψεις και το καθεξής. Θα θέσουν ενδεχομένω και τη θέματα της θεσμικής, των θεσμικών αντιθέσεων και των συνταγματικών αντιθέσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι μια επαναχώρηση σε θέματα κρατού δικαίου δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την ταυτότητα και την πολιτισμική παράδοση, ακόμα και αν διατείνεται κάτι τέτοιο η σχετική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια αυταρχική απόφαση η οποία θέτει σε μειονεκτική θέση την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα θα πρέπει να ε, γίνει μια σαφής διάκριση γιατί η διαφοροποίηση και η ε, ανεκτικότητα αποτελούν όντως ε, ευρωπαϊκές αξίες, αλλά θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε από τις, ευρωπαϊκ... από τις διαφορές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν το ευρωπαϊκό έργο αυτά σε ό,τι αφορά την ανάγκη δημιουργία ενό πίνακα επιδόσεων, ενό scoreboard. Να δούμε τώρα πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο scoreboard. Έχουμε διάφορου ορισμούς σε ό,τι αφορά το scoreboard. Εμεί έχουμε συμπεριλάβει έναν ευρύ ορισμό, ένα συνδυασμό της ε, συζήτησης, αξιολόγησης, ε, ε, ε ορόσημων. Και από την έννοια αυτή το scoreboard θα ήταν μια διαδικασία η οποία θα συμπεριλάμβανε ε, πολλούς φορείς και πολλά στοιχεία. Στην ερευνητική μας ομάδα και μεταξύ των ερωτηθέντων υπήρχε κοινή κατανόηση ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επανεφεύρουμε τον τροχό. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους μηχανισμούς αξιολόγησης και εποπτείας που ήδη υπάρχουν χρησιμοποιούνται επίσης τέτοια μοντέλα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ούτω καθεξής σε άλλους οργανισμούς. Εκ παραλλήλου, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συνένωση δεδομένων από διάφορες πηγές και η ανάλυση τέτοιων συνεργασιών, ακόμα και το να κάνουμε συγκρίσεις, ε, είναι ένα δύνατο σχεδόν εγχείρημα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, διαφορές ε, στη μεθοδολογία και στην ερμηνεία και στη συλλογή των στοιχείων και το καθεξής. Στο επόμενο σημείο θα δείτε ότι όποτε από πλευράς ε, διεθνούς προσκυνίου υπάρχουν ανησυχίες, διατηρούνται τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Δηλαδή, ο μηχανισμός κράτους δικαίου σε καμία περίπτωση δεν θα επεκταθεί σε εξωτερικούς ε, φορείς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει το δικό της σύστημα ε, για να θέσει ενδεχομένω πιο υψηλά πρότυπα από άλλους διεθνούς φορείς. Για να μην είμαστε στο έλεος εξωτερικών οργανώσεων θα μπορούσαμε να έχουμε δικούς μας ε, μηχανισμούς ε, ελέγχου και επιτήρησης και να υπάρξει πρόληψη περιστατικός υπονόμευσης του κράτους δικαίου. το scoreboard θα μπορούσε να ταιριάξει στο χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρθηκε ήδη, και να ενταχθεί στον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης. Ένα από τα βασικά ζητήματα οποιοδήποτε scoreboard είναι το θέμα της νομιμότητάς τους. Ένα αντικειμενικό πλαίσιο είναι απαραίτητο ασφαλώς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ανεξαρτησία και οικονομική αριστεία όλων των συμμετεχόντων. Το επόμενο θέμα που θα εξασφαλίσει την νομιμοποίηση είναι ότι δεν υπάρχουν ε, ορισμοί από τους οποίους που είναι χαραγμένοι στην πέτρα και δεν υπάρχει καμία ιδανική, κανένας ιδανικός τύπος για να πετύχουμε το κράτος ε, δικαίου είναι πολύ ευρύς ο όρος και θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται αναγκαστικά ένα ποσοστό ασάφειας. Τονίζω λοιπόν αυτή την απέτηση να υπάρξει μία ασάφεια για να μην καταντήσει ένας κατάλογος ε, στοιχείων του κράτους δικαίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια γνωστά στοιχεία. Το βασικό θέμα δεν είναι ενδεχομένω ποιοι είναι οι δείκτες, αλλά ποια πρότυπα θα πρέπει να επιλεχθούν, τα οποία να αποτυπώνονται στη συνέχεια από τους δείκτες. Είχε γίνει μία, μάλλον η απόπειρα να δημιουργηθεί ένας κατάλογος στοιχείων, θεωρώ ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο στοιχείο, το οποίο θα συγκεντρώσει τα πειρά της κριτικής για να τονίσουμε λοιπόν πόσο απαραίτητο είναι το στοιχείο της ασάφειας. Συχνά συμβαίνει τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται υπό επιτήρηση να αναφέρουν άλλες, ε, άλλα ε, περιστατικά από γειτονικέ ε, χώρες. Αλλά δεν είναι δυνατόν φυσικά να υπάρξει ένα συγκερασμό των ε, ε, χείριστων πρακτικών, ακόμα και αν όλα τα στοιχεία αυτά όντω υπάρχουν και έχουν εμφανιστεί σε κάποιες άλλες χώρες. Άρα, για να διασφαλίσουμε την νομιμότητα, θα πρέπει να δούμε για ποιους σκοπούς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το scoreboard, ο πίνακας αυτός επιδόσεων. Δεν μπορεί να γίνει κατάταξη, δεν μπορεί να γίνει προστασία κανενός βάσει ε, του scoreboards και δεν μπορεί να γίνουν απλοϊκές ε, αναλύσεις από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση και κατά περίπτωση εξέταση των κρατών μελών ε, λίστα για, ιδιαίτερη για κάθε χώρα για τα βασικά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι η ίση αντιμετώπιση των κρατών μελών. Η χρήση δύο μετρών και σταθμών προφανώς θα αφαιρέσει η νομιμοποίηση οποιοδήποτε τέτοιου scoreboard. Και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω ε, δυσκολίες αν υπάρχουν τέτοια παραπτώματα. και να χρησιμοποιηθεί το διευθυντικό σκέλος του άρθρου 7, όπως είδαμε πρόσφατα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ταχύτητας. Όποιο υψηλή είναι η ποιότητα των δεδομένων, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το scoreboard. Ωστόσο, ε, η ποιότητα φυσικά έχει το τίμημα της σε ό,τι αφορά ε, την ταχύτητα. Δυστυχώς, αν υπάρχει μεγάλη ταχύτητα, ενδεχομένω να προκληθεί ε, ανεπανάρθωτη βλάβη και προφανώς με την παράδοση του χρόνου να χάσει και την αποτελεσματικότητά του ο πίνακα. Αντίθετα, αν είναι υπερβολικά ε, μα, αργή η διαδικασία, ενδεχομένω τα κράτη-μέλη να ισχυριστούν ότι ε, δεν ισχύει η διαδικασία ελέγχου, καθότι δεν ε, είναι σωστά και ακριβή τα στοιχεία. Ας ε, μην χρησιμοποιήσουμε όμως προδιαγραμμένα ε, συστήματα ε, για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων αυτών. Επίσης, πολλές πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από τους εφιστάμενους μηχανισμούς, αλλά ενδεχομένω να χρειαστούν παρόλα αυτά επιπλέον ε, πληροφορίες. Και αυτές μπορούν να συλλεχθούν από, μια ευρεία, από ένα ευρύ φάσμα πηγών τους μη κρατικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, μέσα ενημέρωσης, επίσημες οργανώσεις για την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαμεσολαβητών, εποπτών και ούτω καθεξής. Και φυσικά από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, ομάδα εργασίας του Άρτικου και του καθεξής το Επίσης θα πρέπει να διευκρινίζεται ποιος θα πρέπει να αποδείξει τι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία επαναχώρησης του κράτους ε, Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν συγκεκριμένε κατηγορίε, ε, υπεύθυνο θα είναι το κράτο μέλο να αποδείξει ότι δεν ισχύουν τα όσα του προσάπτουν και ότι πραγματικά τηρεί εις ευρωπαϊκής αξίας. Βλέπουμε λοιπόν τα διάφορα στάδια σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, τρία σενάρια. Στο πρώτο σενάριο τα κρατή-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The member states should, um, uh, should both be scrutinized in order to enhance the legitimacy of... Ε, στο πρώτο σενάριο έχουμε λοιπόν κάνει κάποια σενάρια για να δούμε ποια θα είναι η μεγαλύτερη, ποια θα μπορούσε να έχει την μεγαλύτερη νομιμοποίηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το πρώτο σενάριο δεν έχουμε βασικά προβλήματα για το κατά πόσο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, προβληματικά, μετά έχουμε προβλήματα με διάφορα στοιχεία του κράτους δικαίου. Ας πούμε, μπορούμε, μπορεί να έχουμε μια χώρα που είναι σωστή ως προς το κράτος δικαίου, αλλά, για παράδειγμα, έχει πολύ σημαντικές παραβάσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ας πούμε, στα Ιδρύματα Ψυχικής Υγείας ε, δεν ε, υπάρχουν ε, κατάλληλες συνθήκες. Όλα αυτά, λοιπόν, λαμβάνονται υπόψη για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτίμηση Τη κατάστασης του κράτους δικαίου. Το τρίτο σενάριο όμως είναι ποιοτικό διαφορετικό από το προηγούμενο δύο Να πούμε σε λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε το εγκατάσταση μιας ε, συνδεχματικής ε, κάλυψης μαζί με την έλλειψη παραδοσιακών συστημάτων όπως ας πούμε το διαμεσολαβητή ή ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δύο πρώτα σενάρια έχουμε προωθήσει μια πολιτική ε, λιακάδας ε, <laughs> που έχουμε Ε, έχουμε τα πράγματα, τα, την, την ιδιοποίηση από πλευρά, την οικειοποίηση από πλευρά του κράτου ε, των βασικών θεσμών. Ε, ενώ στο τρίτο σενάριο έχουμε διαφορετική μεθοδολογία και μια δεύτερο, ένα δεύτερο πρόβλημα για τον κύκλο, όπου συστηματικά βλέπουμε πως υποβαθμίζεται η δημοκρατία και γίνονται μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ δεν υπάρχουν λόγοι για να υποθέσουμε τις καλές προθέσεις των όσων ξεκινούν μια τέτοια προσέγγιση, ώστε η ενότητα να επανέλθει στα προβλήματα της κυβέρνησης και μια έννοια που θέλουν να εγκαταλείψει ούτως ή άλλως η εξουσία. Έχουμε λοιπόν διάφορες διαδικασίες, είτε έχουμε το μηχανισμό ή το άρθρο 7 της Ένωσης, το οποίο θα έμπαινε σε εφαρμογή ε, και ο πίνακα επιδόσεων θα οδηγούσε στο να είναι πιο διαφανείς αυτές οι διαδικασίες, ώστε να έχουμε δηλαδή ε, σωστότερες συμφωνίες διοργανικές. Επίσης προτείνουμε μια, τη δημιουργία μιας ε, επιτροπής η οποία θα μπορούσε να επιλεγεί όπως γίνεται τώρα από την Επιτροπή της Βενετίας. Ποια θα έπρεπε να είναι τώρα τα διορθωτικά μέτρα, δεν το έχουμε αυτό εξετάσει στην εκθεσή μας. Πάντως οι προτάσεις μας που προσθέτουν σε αυτή την υπόθεση είναι ε, βασικά το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε με οικονομικές κυρώσεις, ας πούμε παρακράτηση ή μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τώρα μπορεί να είναι παράξενο και αυτές οι κυρώσεις να μην είναι αποτελεσματικές για όλα τα κράτη-μέλη. Για την ώρα είναι ιδιαίτερα ισχυρή τέτοιου είδους ποινές, ε, για οικονομικές ποινές, γιατί παραδόξως ε, οι πρώτες που είναι προβληματικές είναι οι χώρες που είναι και οι μεγαλύτερες ε, δικαιούχοι κοινοτικών χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Λεωνπές από το Πανεπιστήμιο του Μίγκλιστεκ στο Λονδίνο, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση της Εμιλία για τον μηχανισμό δημοκρατίας κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κύριε Πέσ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λοιπόν 10 λεπτά για να παρουσιάσω τα κύρια βρήματα της έκθεσής μας και στην ουσία η αποστολή μας ήταν κάπως διαφορετική. Η έργο μας ήταν να δούμε το γενικότερο πλαίσιο και να εντοπίσουμε τις ελλείψεις προτού διατυπώσουμε προτάσεις, λύσεις και επιλογές. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Στόχος μας λοιπόν ήταν να δούμε τις μικροδιαστάσεις, δηλαδή συγκεκριμένο ε, πεδίο εφαρμογή του δίκτυπη Ωστόσο, θα ήταν ίσως χρήσιμο πριν κάνουμε αυτό να δούμε και κάποιες συστάσεις όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε λοιπόν εάν υπάρχει όντως η αρμοδιότητα παρακολούθησης των κρατών μελών. Αυτό λοιπόν αποτελεί το πρώτο μέρος της έκθεσης όπου ε, απαριθμούμε ορισμένα ζητήματα, εντοπίζουμε δηλαδή ορισμένα ζητήματα και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όντως την αρμοδιότητα παρακολούθησης ε, των κρατών μελών. Έπειτα, όσον αφορά το άρθρο 2, πιστεύουμε ότι ε, η, σημασία και το πεδίο εφαρμογή ε, μπορεί να προκύψει όχι μόνο από την εθνική νομολογία, αλλά και την ευρωπαϊκή. Ως προς αυτό λοιπόν το ερώτημα, εμείς πιστεύουμε πως πράγματι τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, γίνουν αντικείμενο αξιολόγησης για τις συγκεκριμένες αυτές αξίες. σχετικά τώρα με το δεύτερο μέρος της έκθεσης για τα κενά και τις ελλείψεις του φυστάμενου πλαισίου. Καταρχάς είδαμε το πλαίσιο εγκάρσια, δηλαδή εντοπίσαμε τις ελλείψεις από διάφορους τομείς και ίσως η κυριότερη έλλειψη ήταν η διάδοση συγκεκριμένων μέσων και η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, στην ουσία, φάνηκε σαν τα μέσα αυτά να συγκεντρώνονται, να δημιουργείται το ένα μετά το άλλο, να μην υπάρχει όμως κανένας συντονισμός μεταξύ τους και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, θα πούμε ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού οφείλεται στο ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασίζεται στο ότι από τη στιγμή που προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνεσαι και με τις θεμελιώδεις της αξίας. Και αυτό ίσως εξηγεί και τις ελλείψεις που παρατηρούνται, τις εκάρσεις αυτές ελλείψεις που συζητάμε σήμερα. Αυτή η εικασία όμως δεν ισχύει πλέον. Όταν εντοπίσαμε ελλείψεις, εντοπίσαμε ελλείψεις σε συγκεκριμένα μέσα. Δεν θα τις αναφέρω βέβαια εδώ, γιατί η έκθεση είναι αρκετά μεγάλη, όμως αυτό που είδαμε είναι το πλαίσιο κράτους δικαίου, τα νέα μέσα που ε, τέθηκαν σε ισχύ το 2014, τα υφιστάμενα μέσα, αυτό που λέμε nuclear option, δηλαδή ο πυρήνας των επιλογών μας. Επίσης εξετάσαμε το πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέσα, πώς ε, τα αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, ποια περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και ποια είναι τα πρόσθετα μέσα, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός συνεργασίας και ε, ταυτοποίησης. Και τέλος είδαμε το πλαίσιο του κράτους δικαίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2014, αλλά και ο διάλογος που άρχισε τον, ε, τελευταίο, τον Νοέμβριο που μας πέρασε και ήταν πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε στην ε, πρόταση λύσεων για τις ελλείψεις που εντοπίσαμε. Αυτές τις βλέπετε εδώ στο παρόν διάγραμμα. Έχουμε τρεις λοιπόν ε, κάθετες επιλογές και τρεις οριζόντιες. Τι εννοούμε το κάθετες επιλογές. Αυτές είναι δηλαδή λύσεις, επιλογές, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Κατά περίπτωση, γι' αυτό λοιπόν είναι και κάθετες επιλογές. η πρώτη κάθετη επιλογή. Είναι στην ουσία μια επιλογή για την υφιστάμενη διαδικασία επιβολής του νόμου, όπως ε, προβλέπει το άρθρο 258 της Συνθήκης στην την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, δηλαδή να εφαρμοστεί διαφορετικά όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα ε, κατά παραβιάσεων. Θα μπορούμε δηλαδή να εφαρμόζουμε την ε, διαδικασία επιπαραβάση με έναν διαφορετικό τρόπο, σε περιπτώσεις δηλαδή όπου παρατηρούνται κατά συρροή παραβιάσεις που είναι μέρος ενός σχεδίου αποδόμησης του συνταγματικού πλαισίου. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή αφορά μικρές βελτιώσεις στον υφιστάμενο μηχανισμό. Και εδώ εννοώ το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου που εγκρίθηκε το 2014. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες μικρές αλλαγές οι οποίες θεωρούμε πως θα επιφέρουν ασφάλεια δικαίου εφόσον αφορούν το κράτος δικαίου. Θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωση σχετικά με το σύστημα που αξιολογούνται οι απειλές και με την έναρξη χρησιμοποίησης αυτού του πλαισίου. Εδώ να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Τρίτη επιλογή. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους τρόπους χρηματοδότησης ομάδων της κοινωνίας των πολιτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι περισσότερο συνεπής και να κάνει στο εσωτερικό της ό,τι και στο εξωτερικό της. Έχουμε κάνει μια φιλόδοξη πρόταση, ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο όμως, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ίσως μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και πώς μπορούμε να τα ε, ε, χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, το σύστημα χρηματοδότησης Jean Monnet, το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχές, δεν ήταν όμως εύκολο για τις ομάδες κοινωνίας των πολιτών να το χρησιμοποιήσουν και να αντλήσουν κονδύλια από αυτό. Αυτές λοιπόν είναι οι κάθετες επιλογές που έχουμε. Επίσης, έχουμε και ορισμένες οριζόντιες επιλογές. τις οποίες ταξινομήσαμε από την ε, λιγότερο στην περισσότερο φιλόδοξη, απαιτητική αν θέλετε επιλογή. Η λιγότερο απαιτητική νομικά, νομικά όχι πολιτικά επιλογή θα ήταν το να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο έχει, δια, έχει δημιουργήσει τον ε, διάλογο για το κράτος δικαίου. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη διαφάνειας στον διάλογο αυτόν και θεωρούμε πώς θα βελτιωθεί. Έχουμε κάνει και ορισμένες πρόσθετες ε, προτάσεις, όμως το κύριο θέμα είναι η έλλειψη διαφάνειας και ο τρόπος σύστασης του διαλόγου. Δεύτερη οριζόντια επιλογή είναι στην ουσία ένας νέος τύπος συζήτησης που θα συμπεριλάβει τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα συμμετέχουν οι Ευρωβουλευτές και οι Βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων στη συζήτηση για ε, το άρθρο 22. Στην ουσία αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την πρώτη επιλογή, δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Και τέλος, η πιο φιλόδοξη πρόταση που αναφέρεται στην έκθεση είναι αυτό που πρότεινε και ο συνάδελφός μου. Δηλαδή, εμείς τι προτείνουμε, την δημιουργία ενός νέου μόνιμου εγκάρσιου κύκλου παρακολούθησης στον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε τον πίνακα επιδόσεων για τις ε, θεμελιώδεις αξίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα νέο μέσο το οποίο θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη και ενδεχομένως να πρέπει και τα ίδια τα θεσμικά όργανα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λογοδοτήσει για τις ε, πράξεις της. Είναι δηλαδή μια προσθήκη στις αξίες του άρθρου 2. Δεν, είναι δεν πρέπει να είναι κατά ανάγκη ετήσιος ο κύκλος, μπορεί να είναι και εξάμηνος ε, ή μπορεί να μην είναι μόνιμος. Αυτές λοιπόν ήταν οι έξι επιλογές που ε, προτείναμε και με χαρά μου να ακούσω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και σας ευχαριστώ γιατί όλα όσα μας εκθέσατε δείχνουν ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Χρειάζεται να συνεργαστούν πολλοί φορείς και να γίνει και πολύ να δοθεί πολύ ε, δημοσιότητα αλλά και να υπάρξουν πολλές δράσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους ε, θέλει να θέσει ερωτήσεις. Για, διαφορετικά, εγώ θα ήθελα κάτι να πω, διότι συχνά ακούμε αυτή την παρατήρηση για το δίλημα της Κοπεχάγης. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω αν ποτέ κανείς έλεγξε, επί τη βάση ποιων κριτηρίων και μέτρων μπορούμε να ανακαλύψουμε αν υποψήφιο μέλος μπορεί να ακολουθήσει το κράτος δικαίου, μπορεί να ακολουθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα το άρθρο 2, αλλά να ρωτήσουμε το ίδιο για τα κράτη-μέλη πάντοτε ακούμε ναι, όχι, εκεί δεν είναι απαραίτητο να ελέγξουμε. Είτε δεν έχουμε κριτήρια λοιπόν για τα κριτήρια της Κοπεχάγης ή είτε πρόκειται για έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και όταν αναφέρατε τα υφιστάμενα μέτρα, αναφέρατε τον πίνακα επιδόσεων, αλλά όχι τα ίδια τα κριτήρια της Κοπενχάγης και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να βρούμε. Συμφωνώ δε απόλυτα ότι αναφέρατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή όταν μιλάμε για το άρθρο 7 εστιάζουμε στις στους μηχανισμούς κρίσης, ενώ πολλά σπουδαία πράγματα έχουν ήδη γίνει. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ή που θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα είδος μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν κανείς έχει την καλύτερη βούληση, την καλύτερη θέληση, κάποια απόφαση να είναι υπερβολική ή να ακολουθεί λάθος κατεύθυνση και θα μπορούσαμε με φιλικό τρόπο με όλους τους φορείς να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και να αποφύγουμε ένας λανθασμένος τρόπος να καταλήγει τελικά σε κρίση. Είναι καλό να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό και εγκαίρες προειδοποίησεις και να μην μιλάμε ε, για μία κυβέρνηση, για την άλλη κυβέρνηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί για να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αυτά είναι δουλειά που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε. Αν δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο ή να προσθέσει κάτι. I think if there Και αν δεν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις... Α, ναι, με συγχωρείτε. Είστε μπροστά στα μάτια μου και εγώ δεν σας βλέπω. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτών των εισηγήσεων γιατί είναι πολύ σημαντικές. γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα και μπορούμε να δουλέψουμε στο ενέκθεση αυτή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την γραφειοκρατική μας ε, φαντασία και το ευρώ, αλλά ε, να σας πω ότι ε, για την Πολωνία ε, που προέρχομαι και για όλες τις πολιτικές ομάδες και για όλους μας ήταν προφανές ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει σχετίζονται όλα αυτά με την ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εξουσίες και τώρα φάνηκε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας να συνεργαστούμε μαζί όλοι, όχι για να τσακωνόμαστε, όχι για να ε, ε, υπερασπίσουμε τους συμπολίτες μας στη δημοκρατία. Και εντάξει, αυτό μοιάζει με πολιτική δήλωση που λέω τώρα, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουμε αυτό και να προσαρμοστούμε στην πραγματική κατάσταση και την πραγματική δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης στις χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ, Σόφη, για αυτή την, την πρωτοβουλία, γιατί νομίζω πως είναι σημαντική. Στην πρώτη μας συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και αυτή η ιδέα για το σύμφωνο για τη δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο τα θέμα να έχουμε κάποιους μηχανισμούς αξιολόγησης της δημοκρατίας είναι και θέμα του πώς οι χώρες θα ασχοληθούν και οι πολίτες των χωρών σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης της δημοκρατίας τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η κυρία Σόφιντ θέλει να πάρει το λόγο. Δεν έχω ερώτηση να απευθύνω. Γιατί φυσικά ήμουν σε επαφή με τους συντάκτες της ε, έρευνας αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που επισημάνετε κι εσείς, ότι το άρθρο 2 ουσιαστικά είναι το βασικό άρθρο εκείνης της συνθήκης. Το άρθρο 1, όπως λέω, είναι ένας χειρατισμός και το άρθρο 2 περιλαμβάνει την ουσία. Και έχω διαβάσει ό,τι έκθεση έχει περάσει από το χέρι μου και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να βρούμε μια σωστή νομιμική βάση για να εφαρμοστούν οι πρακτικές ε, οι αξίες αυτές στην πράξη. Μια διαθεσμική συμφωνία χρησιμοποιείται ως όρος ή ελλείψη άλλου κατάλληλου όρου. Όπως είπατε και εσείς είναι λίγο ε, το τέρας του Φραγκεστάιν. Να το λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να βρούμε τρόπους ε, να τιμωρήσουμε τις χώρες οι οποίες ε, συμπεριφέρονται λάθος. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα θετικό κύκλο, όπου ως Ευρωπαίοι πολίτε, πολίτες ορίζουμε από κοινού τις αξίες μας. Αυτό κάνει διαφορά και σε βάθος χρόνου. Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, εγώ προσωπικά ε, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να το ορίσει κανεί με μαθηματικού τύπου, σαφέστατα, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια, ε, σε κάποια ορισμένα όρια η δικαιοσύνη, η λειτουργία του ε, δικαστικού σώματος, ε, όλα αυτά είναι σαφή. Μπορεί να αλλάξουν και ασφαλώς και θα πρέπει να αλλάξουν βάσει συζήτηση, αλλά δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο η συνθήκη. Σας ευγνωμονώ ωστόσο για τη δουλειά που κάνατε γιατί κομμάτι-κομμάτι νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε σε ένα πλαίσιο, σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να καταφέρει να λειτουργήσει. Και θα χαρώ ε, να συνεχίσετε να μας διαθέτετε τα στοιχεία σας αυτά. Και είμαι βέβαιη ότι τα αποτελέσματα της ε, μελέτης σας θα δημοσιευθούν και στο, στην σελίδα τη διαδικτυακή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ, Σόφη. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάποιος από τους προσκεκλημένους μας. Εν συντομία, εν συντομία, γιατί ξέχασα να αναφέρω ότι η έκθεση δεν εξέτασε μια λύση ε, που θα συμπεριλάμβανε ε, αναθεώρηση της συνθήκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έλλειψη, σε ό,τι αφορά μηχανισμούς έγκρισης ε, να σας πω ότι έχουμε δύο ουσιαστικά τέτοιου μηχανισμούς, έναν που δεν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε, άρθρο 7 παραγραφός 1, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν υπάρχει υποψία παραβίασης των θεμελιδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε και, και στην συνθήκη του 99. Είναι αυτό ε, κατά μία έννοια ένας ε, μηχανισμός έγκαιρη προειδοποίηση, γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει απαραίτητα ήδη παραβίαση. Και ύστερα είπατε ότι το πλαίσιο κράτους δικαίου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός ε, έγκυρης προειδοποίησης, γιατί ουσιαστικά τη συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων για να διαπιστωθεί κατά το υπάρχει συστηματική παραβίαση του κράτους δικαίου. Άρα έχουμε και δύο, μάλιστα, μηχανισμούς. Τελευταία σχόλια και κλείνω εδώ. Σε ό,τι αφορά τον ασαφή χαρακτήρα του κράτους δικαίου, θα πρέπει να συμφωνήσω με την ε, βουλευτή. Συμφωνούμε. Οι πιο πολλές ε, διεθνείς οργανώσεις έχουν συμφωνήσει επί κάποιων ορισμών ε, λειτουργικών για το κράτος δικαίου και τους χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η συμμόρφωση με το κράτος δικαίου είναι ένα, ένα ζήτημα ποσοστιαίο. Είναι η συμμόρφωση διαρκώς ε, με κάποιες αρχές και ασφαλώς θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση υποθέσεις, κατά πόσον όντως υπάρχει παραβίαση. Εγώ προσωπικά και μιλώ προσωπικά, τον τονίζω αυτό, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι ανοιχτό και ασαφές ο ορισμός δηλαδή του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος και νομίζω ότι πάντα θα είναι μεγάλη πρόκληση αυτή, γιατί ακόμα και με σαφή μέτρα... Α, συγγνώμη, θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Φυσικά και λάβαμε υπόψη τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Φυσικά δεν είχα την ε, δυνατότητα να σας παρουσιάσω στο λίγο χρόνο 80 σελίδες ε, μελέτης. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, με μια πολύ μικρή τροποποίηση, ας μην τα λέμε κριτήρια της Κοπενχάγης για τα μελλοντικά κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ε, όλα τα κρατη πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση. Τώρα, σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούν το κράτος δικαίου, συμφωνώ και εγώ με την εισηγήτρια όλοι αντιλαμβάνονται πότε υπάρχει απόκληση από το κρατός δικαίου. Ωστόσο, υπάρχουν και διαβαθμίσεις και υπάρχουν επίσης και πάρα πολλοί ε, χρήσιμοι δείκτες. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν κατάλογο με ε, δείκτες ή με ε, υποδιαιρέσεις του κράτους δικαίου. Και πιστεύω πως η κυρία Ιντφέλντ ως εισηγήτρια αναγνωρίζει την έμφαση που πρέπει να δοθεί στους ε, δείκτες ε, ποιότητας ε, και την αξιολόγηση κατά περίπτωση στα κράτη-μέλη κατά τον έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μας δείχνετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην δική μας έκθεση και πιστεύω πως θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψε τους επόμενους μήνες για το θέμα αυτό εδώ. Και ελπίζω ακόμα και με το Συμβούλιο. Έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην ε, απόφαση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και ελπίζω να συνεχιστεί η καλή μας συνεργασία. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο προβλέπεται για τις τέσσερις και ενδεχομένως ορισμένοι συνάδελφοι να μην έχουν έρθει έως τότε. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να διακόψουμε την συνεδρίαση και θα σας δείσω να επιστρέψετε στις τέσσερις ακριβώς. Κάντε ένα διάλειμμα για καφέ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της απογευματινής μας ημερησίας διάταξης, η πώληση ηθαγένεια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταγγελίες για διαφθορά στην έκδοση τίτλων διαμονής και θεωρήσεων από προξενία και πρεσβείες κρατών μελών σε τρίτες χώρες και πιθανότατες συνέπειες για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη σε σχέση με την πώληση ηθαγένειας έχει γύρει ανησυχίες ανάμεσα σε ορισμένα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Γι' αυτό και οι συντονιστές αποφάσισαν να θέσουν το θέμα αυτό υπό συζήτηση και καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ενημερώσει σχετικά με το τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το ζήτημα αυτό. Έπειτα, όσα μέλη θέλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση θα λάβουν το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Δημητρακόπουλο και τον Κυρία Δημητρακόπουλο, έχετε το λόγο. Thank you, um, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την ε, κυρία Δημήτρη Κοπούλη, ονομάζομαι Χίλμουτ και είμαι από το ίδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνοδεύομαι από τον ε, συνάδελφο τη ΓΑΜΑ που θα σα ε, μιλήσει περισσότερο για ζητήματα ασφαλεία σχετικά με την πώληση ηθαγένεια όπως επιβεβαίωσε και το δικαστήριο στην ομολογία στην υπόθεση Walkman, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ε, θέσει τους κανόνες για την απόκριση και απώλεια ηθαγένειας. Όμως, την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την το ευρωπαϊκό δίκαιο. η χορήγηση ηθαγένειας ενός κράτους μέλους έχει και ε, διάφορα προελκόμενα, όπως για παράδειγμα ελεύθερη μετακίνηση, ε, δικαίωμα εγκατάστασης, εκλέγην και εκλέγεστε στις ε, δημοτικές εκλογές της χώρας κατοικίας και απόκτηση υπηκότητας. Δεν είναι λοιπόν μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα κράτος μέλο και ενώ γίνεται σεβαστή η αυτονομία των κρατών μελών, είναι ωστόσο καθήκον μας να ε, προστατεύσουμε το, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ε, εξουσία αυτή, καλή την πίστη και με καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις αλλά και το διεθνές δίκαιο και τα κριτήρια πάνω στα ε, οποία βασίζεται η εθνική νομοθεσία. Τα κριτήρια αυτά απαιτούν την ύπαρξη ενός ε, συνδέσμου ανάμεσα σε, αυτόν που αιτείται την ε, ηθαγένεια και στην χώρα ε, που θα του χορηγήσει την ηθαγένεια. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει αναλύσεις σχετικά με διάφορα σχέδια επενδυτών ε, που αποκτούν ηθαγένεια. Υπάρχουν κρατημέλη δηλαδή τα οποία χορηγούν ηθαγένεια και όχι απλά κατοικία σε ορισμένους επενδυτές ή ορισμένε συνθήκες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο σύνδεσμος αυτός, η ύπαρξη συνδέσμου ανάμεσα στο άτομο και στο κράτος μέλους. Η Μάλτα τροποποίησε την νομοθεσία της για να αλλάξει η απέτηση κατοικίας πάνω από, σε, σε τουλάχιστον μάλλον 12 μήνες στη χώρα υπάρχουν διάφορα άλλα τέτοια σχέδια ε, επενδυτών εντό εισαγωγικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή γίνεται διάλογος με ένα κράτος μέλος το οποίο δίνει την ε, ηθαγένεια μόνο ε, μετά από κάποια επενδυτική πρωτοβουλία, η Κύπρος δηλαδή. Έχουν γίνει πολλές ανταλλαγές απόψεων, πολλές συναντήσεις ανάμεσα στις Κυπριακές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 2014 και 2015. Και με βάση το αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, αναλογιστεί το ε, ποια δράση θα αναλάβει. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτά τα σχέδια απόκτηση ηθαγένεια σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και θα ενημερώνουμε την Επιτροπή όταν ε, αυτό είναι αναγκαίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ε, DG Home θα αναφερθώ στη δεύτερη πτυχή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια για την χορήγηση ε, ε, τίτλων διαμονή, ή χρυσών θεωρήσεων όπω ονομάζονται. Αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Για να είμαστε σαφεί, αυτέ οι χρυσέ βίζε είναι άδειε παραμονή, όχι για διαμονή στη Σέγγεν. Αυτές οι, η έκδοση τέτοιων θεωρήσεων εναντί επενδύσεων δεν είναι αρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη ορίζουν τους όρους για την είσοδο και διαμονή των ε, πολιτών τρίτων φορών που θέλουν να επενδύσουν και να μείνουν πάνω από τρεις μήνες. Ωστόσο, οι δικλείδες ασφαλείες που υπάρχουν για τις, ε, τα σύντομα ταξίδια έχουν να κάνουν με την ε, ζώνη και γενικά εθνική, ε, εθνικός τίτλος διαμονής δεν έχει να κάνει με την διαμονή στο εσωτερικό. Και όσοι έχουν τέτοιους τίτλους δικαιούνται για να ταξιδεύουν έως 90 ημέρες σε άλλα κράτη Σέγγεν και θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους εισαγωγής για όλα τα κράτη. Αν ε, ένας επίκος χώρας δεν πληρεί τους όρους αυτούς σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, νόμιμα το κράτος μέλος που έχει εκδώσει την αντιδιαμονή σε, θα πρέπει να δεχτεί το άτομο αυτό στην επικρατεία του και πάλι. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αρνηθούν την είσοδο στην επικράτειά τους ή να διώξουν υπηκόου τρίτος χωρών που αποτελούν σοβαρή απειλή στη δημόσια ασφάλεια της χώρας. Σε ό,τι αφορά τη μακρά παραμονή σε άλλα κράτη-μέλη, οι εθνικές άδειες διαμονή σε ένα κράτο μέρο δεν συνεπάγονται αυτόματα δικαίωμα διαμονή σε άλλο κράτο. Μόνο όσοι έχουν θεώρηση βάσει τη ε, θεώρηση τη οδηγίε για τι ε, μακροπρόθεσμε ευρωπαϊκέ θεωρήσει έχουν τέτοιο δικαίωμα. Να σα διευκρινίσω ότι αυτέ οι μακροπρόθεσμες άντρε παραμονή δεν έχουν να κάνουν με τι εθνικές άντρε παραμονή. Οι άντρε παραμονή τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χορηγηθούν μόνο βάσει των όρων που ορίζονται στη σχετική οδηγία και είναι πολύ αυστηρή η σχετική όρη, για παράδειγμα, διαρκής παραμονή στη χώρα τουλάχιστον πέντε έτη, επί πέντε έτη. Και τώρα να στραφώ σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί την επιστροπή σας. Ε, ενδεχόμενη σε σύνδεση με τη διαφθορά και σε ό,τι αφορά τι επενδύσει και καταγγελίε περί διαφθορά στην έκδοση τη διαμονή και θεωρήσεων από προξενία και πρεσβείε. Η πρόληψη τη ε, διαφθορά αποτελεί προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολουθούμε λοιπόν την ακεράτητα των κρατών μελών και τις πολιτικές κατά της διαφθοράς μέσω σχετικών μελετών και ερευνών. Το 2014 δημοσιεύτηκε μια τέτοια πρώτη α, μελέτη. Τα βασικά α, μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο κατά περίπτωση και μέτρα τα οποία υποστηρίζονται από ευρωπαϊκού πόρου. Όπου υπάρχουν κατηγορίε διαφθορά, οι εθνικέ αρχέ είναι αυτέ που πρέπει να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν ενδεχόμενη απάτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει γιατί πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα η έκδοση τέτοιων τίτλων. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουν οδηγήσει τέτοιε έρευνε σε μεταρρύθμιση τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, μετά το σκάνδαλο του 2014 με τι χρυσέ θεωρήσει που οδήγησε και σε παρέτηση του Υπουργού Ιστορικών. Ωστόσο, η διαφθορά υπονομεύει το κρατό δικαίου, την νομιμότητα των ε, θεσμικών οργάνων και ενδεχομένω και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών σε περιπτώσει διαφθορά σε ό,τι αφορά την χορήγηση βραχυπρόθεσμη θεώρηση, υπονομεύει και το Σένιεν. Η καταπολέμηση λοιπόν της διαφθοράς είναι σημαντικό τμήμα του θέματο που τίθεται. Πρωτού εκδοθεί λοιπόν ένα εθνικό τίτλο διαμονή, το κράτο μέλο θα πρέπει να, διαβου... να συμβουλεύεται το ΣΥΣ. Δεν θα πρέπει να χορηγείται λοιπόν τέτοιο τίτλο σε ένα άτομο για το οποίο υπάρξει... υπάρχει σήμα στο ΣΥΣ. Επιπλέον, επειδή πρόκειται για επενδύσει, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματο ε, εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που κάνουν τέτοιε επενδύσει. Επιπλέον, οι εθνικέ πολιτικέ κατά τη διαφθορά υποστηρίζονται και παρακολουθούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σχετικά εργαλεία. Η Κομισιόν παρακολουθεί λοιπόν την ακαιρεότητα των κρατών μελών μέσω των σχετικών ερευνών, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι κατά τη διαφθοράς και τα ευρωπαϊκά σημεία επαφής και τα ευρωπαϊκά δίκτυα κατά τη διαφθορά, αποτελούν πλατφόρμες κατά τη ε, διαφθορά και για τη συνεργασία των αρχών για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη διαφθορά. Ανταλλάσσουν λοιπόν ε, εμπειρίε και πληροφορίε, ε, διασυνοριακά, αναπτύσσουν κοινέ στρατηγικέ και θέτουν υψηλά πρότυπα και κάνουν συστάσει σε αλλήλους. Επίσης, ε, δημοσιεύτηκε ένα εγχειρίδιο για την αυτοαξιολόγηση των ε, αρχών επιβολής του νόμου για την ε, μεγαλύτερη ακαιρεότητα. Επίσης, υπάρχουν και μέθοδοι καταπολέμησης της διαφθοράς σε ό,τι αφορά τους συνοριακούς ελέγχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Λίκη και Πρόεδρος. σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στις διαφορές ανάμεσα στην ηθαγένεια και την ε, θεώρηση παραμονής ε, ή την χρυσή θεώρηση. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή που δέχτηκε την πρόσκλησή μας για τη σημερινή αυτή συζήτηση γιατί μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το διακύβευμα εδώ είναι πολύ σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο. Η πώληση της ηθαγένειας είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια επιφέρει διάφορα δικαιώματα τα οποία ποτέ θα έπρεπε να είναι αντικείμενο πώλησης. Είναι βέβαια κρατική αρμοδιότητα, αλλά είναι και είσοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το μέγεθο του τραπεζικού σου λογαριασμού αν θα πάρει θεώρηση ή όχι. Το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια είναι πολύ αμφίβολο για αυτά τα θέματα γιατί δημιουργούνται πολλά παραθυράκια ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Ε, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μια τέτοια επιλογή. Η έλλειψη σαφήνεια σε σχέση με τα ονόματα των όσων αγοράζουν την Ιθαγένεια, και εδώ μιλάω για τη δίδια μου τη χώρα, τη Μάλτα, αυτό μόνο τονίζει τις ανησυχίες αυτές. Σύμφωνα με τον εθνικό μας νόμο, η ηθαγένεια θα πρέπει να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει γνήσια σύνδεση με τη χώρα. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι εξής. Η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη που ο κόσμος αγοράζει διαβατήρια και μπορεί να ε, έχει πραγματική σύνδεση και σχέση με την ε, ε, κάστοτε χώρα. Σύμφωνα με το, την δική μας νομοθεσία θα έπρεπε να υπάρχει και μια συγκεκριμένη διάρκεια παραμονής. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά κατοικούν σε αυτήν την χώρα, στην κάστοτε χώρα. Για το θέμα της ασφάλειας η Κομισιόν έχει οποιαδήποτε εποπτεία για το τι γίνεται όντως έλεγχος, γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται και αυτό συνδέεται με τη δεύτερο μιλητή, εκπρόσωπο της Κομισιόν που αναφέρθηκε στην διαφθορά. Και όπως είδαμε και με το σκάνδαλο των χαρτιών των εγγράφων του Παναμά, δεν μπορούμε να περιμένουμε να, να, να δεχόμαστε την κατάχρηση των συστημάτων και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ε, ρήτρε ασφαλείας. Και φυσικά αυτό αναφέρεται στην αρνητική προσοχή που δίνεται ε, στην κυβέρνηση της Μάλτας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ Ρομπέρτα ή Μύρια. Ευχαριστώ Μπρίγκετ και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα για το οποίο συζητάμε, γιατί ναι, συμφωνούμε, πώληση της ηθαγένειας χωρίς καμία σχέση με την εκάστοτε χώρα είναι ανησυχητική υπόθεση. Και όπως είπε και ο ίδιος Επίτροπος, το βασικό θέμα που συζητάμε εδώ είναι όχι το να γίνει κυνηγή μαγισσών ενάντια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, γιατί αν δούμε τα διάφορα ε, προγράμματα και διαδικασίες στα διάφορα κράτη-μέλη είναι πολλά και ποικίλα και το έχει αναφέρει και η ίδια η Κομισιόν. Και ως προς αυτό ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν για το κατά πόσο μιλάμε και για το πρόγραμμα μεμονωμένων επενδυτών της Μάλτας. Ε, πρόκειται για ένα ε, κοινό ανακοινωθέν τύπου από πλευρά της Κομισιόν το 2014 που λεγόταν ότι οι τροπολογίε που εισήχθησαν συμπεριλάμβαναν τι γνήσιε σχέσεις και δεσμού με την Μάλτα πριν να υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει κανείς την ε, ε, ηθαγένεια της ε, χώρας. Τότε η Κομισιόν περιέγραψε ότι όλα αυτά γίνονται καλή τυπίστη πίστη και στο πνεύμα συνεργασία. Τόσο μάλιστα που εξέφρασαν την ικανοποίησή του, ε, εξέφρασε μάλλον την ικανοποίησή τη η Προεδρία για την ε, σύμπνοια. Ε, Εμεί από ό,τι καταλάβαμε σήμερα είναι ικανοποιημένη με αυτή την γενική διάταξη. Καταλαβαίνω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις με την Κύπρο σε σχέση με το δικό τους πρόγραμμα, το οποίο μέχρι τώρα σημαίνει ότι μια τρίμηνη περίοδος χορηγείται από την Κύπρο για τους ανθρώπους που δεν είναι πολίτες της Ένωσης, ώστε να τους χορηγηθεί η θαγένεια Πού έχουν φτάσει οι συζητήσει και ποιε περαιτέρω δράση θα αναλάβει η Κομισιόν ω προς αυτό. Η Κομισιόν επίσης δηλώνει πως εξετάζονται και άλλα προγράμματα. Ποια είναι αυτά σε σχέση με τις ανησυχίες για την ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο να προβαίνει κανείς σε ισχυρισμούς για διαφθορά, αλλά η Κομισιόν μας είπε ότι αναλύει την κατάσταση και ότι οποιαδήποτε ισχυρισμοί ή περί διαφθοράς αναλύονται από την ίδια την Κομισιόν. Και επίσης η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η Ιντερπόλ και το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν γνωρίζουν πότε εκδίδεται η θεώρηση και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να προσθέσω μια ακόμη ερώτηση. Ακόμα και αν μόλις ακούσαμε τις διαφορές ανάμεσα στο να έχει άμεσα κανείς την ηθαγένεια ή να πληρώνει για μια χρυσή θεώρηση, καταλαβαίνω ότι εφόσον δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή θεώρηση δεν έχουμε δικαίωμα να το ελέγξουμε αυτό. Η Κομισιόν δηλαδή αναφερόταν βασικά σε ισχυρισμού ευθορά, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ανάλυση σχέση με ένα άλλο θέμα που συζητάμε εδώ και μήνε. Έχοντας υπόψη τα θέματα της μετανάστευσης, δουλεύουμε για να πούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε ποιοι έρχονται στις χώρες μας. Ως προς αυτό λοιπόν, ακόμα και αν είναι μόνο μια εθνική θεώρηση και εθνική ηθαγένεια και στις δύο περιπτώσεις πιστεύω πως είναι δυνατόν για όσους το έχουν πληρώσει να μπορούν να υπάρξουν, να, να μπορούν να δράσουν και σε άλλες χώρες, αλλά το να ή το να κάνουν δουλειές και επιχειρήσει, αλλά κάποιες συμπεριφορέ μπορεί να επηρεάζουν και άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει δηλαδή να ελέγχεται κατά πόσο οι υποψήφοι αυτοί για θεώρηση ε, τηρούν τους όρους για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις. Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την πώληση ηθαγένειας. Είπα ότι ερευνούμε στην παρούσα φάση και ε, διεξαγάγουμε διάλογο με ένα κράτος μέλος, την Κύπρο συγκεκριμένα, για τα άλλα κράτη-μέλη. Ε, παρακολουθούμε την κατάσταση και ενημερωνόμαστε. Εξ όσων γνωρίζουμε όμως, ένα κράτος μέλος, όπως είπα ε, και πριν, χορηγεί πολιτογράφηση μόνο με επενδύσεις στην Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τώρα του κατά πόσον η η είναι όντως, τρίτων ε, χωρών όντω διαμένουν στη χώρα και πραγματικά κατά πόσον υπάρχει ειλικρινή σύνδεσμος μεταξύ του Ετούντα και της χώρας. Οι Μαλτέζικες αρχές είναι αυτές που ελέγχουν στα πλαίσια της δέουσης επιμέλειας κατά πόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμπεριλαμβάνει α, τιμολόγια, λογαριασμού τηλεφώνου, συμμετοχές σε τοπικέ λέσχες, εγγραφή σε σχολεία κτλ. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, το αξιολογούν και το καθορίζουν κατά περίπτωση οι εθνικές αρχές. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση και τη δέσο επιμέλεια και τους ελέγχους στην περίπτωση της Μάλτας θα πρέπει να σας παραπέμψω στους συναδέλφους μου. Θα επανέλθω αν θέλετε στο θέμα αυτό. Οι ανησυχίες ως προς την ασφάλεια για την Interpol, το ε, σύστημα ΒΙΣ, όλα αυτά τηρούνται. Το ΒΙΣ για τους τίτλους διαμονής θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Δεν μπορεί να χορηγείται λοιπόν τέτοια, τέτοιος τίτλος διαμονής σε επικόστο της χώρας. Αν υπάρχει σήμανση του ατόμου αυτού στο ΣΥΣ. Μπορώ να συμβουλευτώ τους συναδέλφους μου για το κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι όροι και να σας ε, ενημερώσω. κατά πόσον υπάρχουν τώρα περιπτώσεις ε, διαφθοράς ε, και επιχειρηματικών πρακτικών ε, που μπορεί να επηρεάσουν και άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ΣΥΣ είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ακολουθούμε ως βάση. Και αυτά, μόνο αυτό μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. I'm so sorry. Um, as no, again... Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε και ερωτήσεις από τους συναδέλφους στην συνέχεια. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και ελπίζω να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον για να μας ενημερώσετε για αυτήν την πρακτική της χρυσή βίζα, όπως ονομάζεται. Νομίζω όμως πως αν δεν υπάρχει κάτι άλλο θα ε, κλείσω τη συνεδρίαση. Προτού όμως φύγετε όλοι, η Μίρια Ντάλη δεν ήθελε να επανέλθει. Ε, Μία ερώτηση πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι διερευνά αυτή τη στιγμή διάφορα περιστατικά, διάφορα τέτοια προγράμματα και θα ήθελα να μάθω τι ε, ακριβώς ερευνά και ποιες χώρες αφορά. Μάλιστα, σε επανέλθουμε λοιπόν στο ερώτημα αυτό. Ποιες είναι οι άλλες χώρες οι οποίες ε, έχουν παρόμοια προγράμματα και ε, τι περιπτώσεις εξετάζετε. Μπορείτε να μας ε, απαντήσετε ή τουλάχιστον γραπτός. Όπως είπα και πριν, δεν διεξάγουμε έρευνες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε μια αξιολόγηση της ε, κατάστασης σε ένα κράτος μέλος. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν έχουν ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό της Κύπρου, ε, τα παρακολουθούμε, είμαστε ενήμεροι και εάν φυσικά παρουσιαστούν αμφιβολίες ή διαπιστώσουμε κάτι, δεν θα διστάσουμε να ανοίξουμε διάλογο με το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε αυτό το στάδιο όμως δεν έχουμε κάποια ένδειξη ε, του ότι θα χρειαστούν περισσότερες ενέργειες από μέρους μας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες και τώρα θα, θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα το απόγευμα και ε, θα λήξει η συνεδρίαση. Μην ξεχνάσετε ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι στο Στρασβούργο τη Δευτέρα το βράδυ στις 7.